Hello and uh, Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο εργαστήριό μας, την ομάδα εργασίας 2. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, αγαπητά μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητοί καλεσμένοι, φίλοι και συνάδελφοι, χαίρομαι ε, που σας καλωσορίζω σήμερα στο δεύτερο workshop που οργανώνουμε με θέμα το φύλλο και την υγειονομική περίθαλψη. Όπως ξέρετε, βιώνουμε ένα τεράστιο κύμα προσφύγων και μεταναστών που προσπαθούν να γλιτώσουν από μαζικές δολοφονίες, ε, πολέμους, διώξεις ε, και βία λόγω φύλου. Οι, πιο ευάλωτοι πρόσφυγες είναι γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες τους, γυναίκες με παιδιά, εγγύες γυναίκες ε, που θυλάζουν, ασυνόδευτοι ανήλικοι, παιδιά με άνθρωποι με αναπηρίες και ηλικιωμένοι. Αυτοί είναι οι πιο ευάλωτοι και έχουν ε, φοβερές ανάγκες που χρήζουν αντιμετώπιση ε, στους καταβλισμούς υποδοχής και διέλευσης, ενώ περιμένουν να διεκπαιρεωθούν οι αιτήσει τους για άσυλο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκες και άμεσες και πιο μακροχρόνιες και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών σε αυτό το πλαίσιο. Δεν θέλω φυσικά να προεξοφλήσω τη συζήτηση ή να προδικάσω τα επιχειρήματα των καλεσμένων και εμπειρογνωμόνων μας και θα ήθελα να περάσουμε αμέσως χωρίς άλλη καθυστέρηση στους καλεσμένους μας. Η πρώτη είναι η κυρία Βιρζίνια Λάγκμπαρκ Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Η οργάνωση αυτή ε, συνδιοργάνωσε αυτό το εργαστήριο και συνέβαλε τα μάλα στο έργο της Επιτροπής Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί Εθνικοί Βουλευτέ, συνάδελφοι, Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες ενός πρωτοφανούς φαινομένου που δημιουργεί τεράστιες πιέσεις στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να περιθάλψουν τους όλο και μεγαλύτερους αριθμούς προσφύγων και ετούν τον άσυλο που παίρνουν τα σύνορα προσβλέποντας ένα καλύτερο μέλλον. Ήμασταν προετοίμαστοι για μια τέτοια κατάσταση. Οι διεθνείς οργανώσεις και εθελοντές ε, συστηματικά μας ενημερώνουν για την έλλειψη του στοιχειωδών ε, στην αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών και της ανάγκης ε, άμεσης ε, παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Στην κατάσταση αυτή ε, είναι δύσκολο να μην ζητούμε όλο και περισσότερες δράσεις. το ταξίδι των, των προσφύγων και του τον άσυλο προς την Ευρώπη είναι επικίνδυνο και γι' αυτό θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματά του και ιδιαίτερα στα προβλήματα των γυναικών και των κοριτσιών. Πρώτα απ' όλα λόγω του φίλου τους. Ε, γυναίκες πρόσφυγες και του εσάσυλο είναι εκτεθειμένες σε ε, ειδικού κινδύνους ε, υγεία, όπω η βία λόγω του φύλου, περιπλοκές στην αναπαραγωγική τους υγεία. Χρειάζομαστε λοιπόν υπηρεσίες που θα λαμβάνουν υπόψη την, την ιδιαιτερότητα του φύλου και θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών και κοριτσιών. Μάλιστα έχουμε σχετικά μεγάλο αριθμό εγγύων γυναικών προσφύγων. Οι περισσότερες μάλιστα υπέστησαν μεγάλο ψυχολογικό στρες και σωματικά προβλήματα. Γι' αυτό και είτε έχουν προώρους στο είτε έχουν επιπλοκές στο τοκετό ακόμη και πρόωρου θανάτου. Έχουμε και πολλές γυναίκες που θυλάζουν και που λόγω του υποσυτισμού αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας, και, ίδιες και τα παιδιά τους. Όλο και περισσότερος αριθμός γυναικών και κοριτσιών μεταξύ των προσφύγων καθιστά επιτακτική ανάγκη την προσαρμογή των εγκαταστάσεων στέγασης και υποδοχής. Το τελευταίο καιρό οι γυναίκε και τα κορίτσια είναι το 60% του συνολικού αριθμού των προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη. Είναι οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι, γυναίκε και τα κορίτσια, χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία, ιδιαίτερα όταν ε, ταξιδεύουν μόνε του, όταν έγκυε ε, θυλάζουν ή όταν είναι ασυνόδευτοι, ανήλικοι, ανάπηροι ή ηλικιωμένοι. Το σύστημα ε, προστασίας μας θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιάζουσες ανάγκες αυτών των πιο ευάλωτων ομάδων. Είχαμε ιδιαίτερε περιπτώσεις ε, ε, προβλημάτων υγείας των γυναικών που επιχειρούν αυτό τον επικίνδυνο διάπλου προς την Ευρώπη. Θα ήθελα να τονίσω κάποια στοιχεία που κατά τη γνώμη μου χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή. Οι γυναίκε και, τα, και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένε στη βία λόγω οι γυναίκες και τα κορίτσια, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουν μόνες τους, είναι πολύ πιο ευάλωτα θύματα ε, βίας, ελαφροδιακίνησης, ε, ε, σωματεμπορίας και επίσης ε, σε πολύ συνοστισμένους ε, χώρους, ε, χωρίς ιδιαίτερους χώρους για τις γυναίκες, είναι πολύ πιο εκτεθειμένες σε σεξουαλική και άλλη παρενόχληση. Χρειαζόμαστε ασφαλείς χώρους στα κέντρα υποδοχής και στέγασης για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Ιδιαίτερους χώρους να μπορούν να θυλάζουν και να χρειάζονται κάποια ιδιωτικότητα για τις υγειονομικές τους ανάγκες. Χρειαζόμαστε περισσότερες νοσηλεύτριες και γυναίκες γυναικολόγους και προσωπικό που θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη διάσταση του φύλου και θα μπορεί να προσφέρει η υγειονομική περίθαλψη και ψυχολογική στήριξη. Επίσης, καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Οι γυναίκες πρόσφυγες και τα κορίτσια πολλές φορές ε, δεν έχουν πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, ε, στους καταβλισμούς διέλευσης ε, ή και στα κέντρα υποδοχής δεν έχουν καλή ενημέρωση, δεν υπάρχουν γυναίκες διερμηνείς. Αυτό αποθαρρύνει τις γυναίκες από το να ζητήσουν βοήθεια, καθιστώντας τις ακόμη πιο ευάλωτες στους λαθροδιακινητές και άλλους καιροσκόπους. Χρειαζόμαστε και περισσότερες γυναίκες διερμηνείς για να εξασφαλίσουμε ενημέρωση ε, των γυναικών και των κοριτσιών για τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται και στις οποίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση. Επίσης, ε, θα πρέπει σε ξεχωριστούς χώρους να γίνονται ιατρική έλεγχοι για να αισθάνονται ασφάλεια γυναίκες κατά κόρηση και να μπορούν να υποφεληθούν από αυτή τη βοήθεια. Αυτά είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα των επιτακτικών αναγκών που χρειάζονται πρόθεσμα. Φυσικά θα χρειαστούν και μακροπρόθεσμες τέτοιες υπηρεσίες μετά την ε, εγκατάσταση αυτών των προσφύγων γυναικών και κοριτσιών. Και οι γυναίκες μετανάστριες ε, ε, προσκρούσε πολλού φραγμού ό,τι αφορά την πρόσβαση σε πιο μακροπρόθεσμε υπηρεσίε υγειονομική προήθαψη. Μερικέ φορέ έχουν ε, προβλήματα και γλωσσικά που του εμποδίζουν να έχουν πρόσβαση. Ή ε, ιδεολογικά, γιατί ε, λόγω των παραδόσεων πολλές γυναίκες, ε, σε πολλές γυναίκες δεν επιτρέπεται να ε, ζητήσουν τη βοήθεια άνδρα γιατρού. Επίσης, ε, πολλές φορές δεν υπάρχουν υπηρεσίες υγείας κοντά στα κέντρα ε, στέγασης, και υποδοχής, οπότε οι γυναίκες δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους. Οπότε οι γυναίκες ε, αναγκάζονται να ζητήσουν βοήθεια μόνο στις ε, έκτακτες και πολύ σοβαρές περιστάσεις. Οπότε ε, οι γυναίκες που εισέρχοντας πρόσφυγες ή μετανάστες στην Ευρώπη, ανά πάση στιγμή μπορούν να, να υποπέσουν σε μια κατάσταση παράτυπη, κάτι που θα καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την πρόσβασή τους ε, στις υπηρεσίες υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιες ε, πρακτικές λύσεις για να βελτιώσουμε την κατάσταση της υγείας των γυναικών ε, προσφύγων και του ανάσυλων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ, η κυρία Λάγκπερ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στη δεύτερη προσκεκλημένη μας, την καθηγήτρια Χάνα Μπρόντε. Αυτή τη στιγμή διδάσκει στο τμήμα κοινολογίας του Πανεπιστημίου της Ουψάλα στη Σουηδία και ερευνά τις σχέσεις μεταξύ υγείας, ρατσισμού και εθνότητας. Ε, έχει δημοσιευθεί στο Sociology of Health and Illness, στο Health and Science και σε ε, στο Sociological Research διαδικτυακά. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω εδώ ενώπιόν σας. Ε, αναφέρομαι κυρίως ε, σε έρευνα ε, την οποία αναλάβαμε για την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το τμήμα της Ευρώπης και εξετάζει τα ερευνητικά στοιχεία σε πολιτικές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για πρόσφυγες και αιτούντες ε, άσυλο. Σε αντίθεση με την πολύ ισχυρή δεντεολογική και νομική σκοπιά της παροχής ε, υγειονομικής περίθαλψης. Ε, ε, τα στοιχεία που έχουμε από πλευράς έρευνας είναι κατακαιρματισμένα, στην καλύτερη περίπτωση. Ε, καταρχάς υπάρχουν ορισμοί πολύ ασυνεπείς και για τους ίδιους τους μετανάστες. Και αυτό φυσικά γίνεται διότι πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία το κατά πόσον κάποιος θα θεωρηθεί πρόσφυγας, μετανάστης ή παράτυπος μετανάστης και είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση που αλλάζει ε, και κατά τη διέλευση συνόρων και ε, για διάφορους άλλους λόγους που δεν μπορούν να ελέγξουν φυσικά οι ίδιοι μετανάστες. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι κατακαιρματισμένα που βασίζεται σε κάποιες ακαδημαϊκές έρευνες και σε στοιχεία από μη κυβερνητικές οργανώσεις, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σοβαρή ανάγκη για υγειονομική περίθαλψη σε εγγύους και θέματα μητρότητας και υπάρχει και πολύ μεγάλη ανάγκη για ε, ψυχικές νόσους και ψυχική αναστάτωση. Ε, υπάρχουν κάποιες έρευνες και βλέπουμε ότι έχουν πενταπλασιαστεί τα ποσοστά. Ε, Υπάρχει επίσης και πολύ μεγάλη ανάγκη για πάρα πολλές ε, παθήσεις οι οποίες δεν έχουν ε, ε, καταγραφεί και δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Ένας άλλος τομέας ο οποίος απασχολεί την έρευνα τακτικά είναι θέματα επικοινωνίας και γλώσσας, τα οποία ήδη ακούσαμε. Ε, που σίγουρα ε, αποτελούν πρόσκομα για την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, αλλά δεν είναι μόνο γλωσσικό πρόβλημα, είναι και θέμα προσδοκιών, ε, αντίληψης, αβεβαιότητας και φυσικά έλλειψης εμπιστοσύνης. Δεν είναι μόνο θέμα ύπαρξης διερμηνίας για να υπάρχει πρόσβαση ότι αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε στην έρευνα έχουμε πολύ λίγες ιστορίες από τους ίδιους τους πρόσφυγες. Οι έρευνες συνήθως δίνουν στοιχεία για τις απόψεις επαγγελματιών, αλλά ε, φωνές ε, γυναικών προσφύγων είναι σπάνιες και συνήθως ο ορισμός που δίνουν για την υγεία είναι ολιστικός δεν θέλουν απλώς αντιβιωτικά, θέλουν ένα πλαίσιο ε, στο οποίο να μπορέσουν να ζητήσουν υγειονομική περίθαλψη και αυτά είναι τα θέματα που τους απασχολούν. Ένα από τα πράγματα λοιπόν τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε σαφέστατα από τα ερευνητικά στοιχεία είναι ότι ε, πράγματι το νομικό πλαίσιο που διέπει τη μετανάστευση είναι αυτό το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Το γεγονός ότι κρατούνται, ότι τους εκτοπίζουν και η όλη φύση και η διάρκεια της διαδικασίας αίτησης ασύλου δημιουργούν και αυτά προβλήματα υγείας. Γραφειοκρατικό κόστος, κόστος γενικότερα, άλλη φραγμή κυρίως όσον αφορά τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και αυτά δημιουργούν προβλήματα υγείας. Και επικρατεί κάπως η υπόθεση που θα θίξει και η συνάδελφος ότι συνήθως η τραυματική κατάσταση που βιώνουν πριν φτάσουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές που δημιουργούν τα προβλήματα και θεωρούνται ότι αυτά όλα θυσορεύονται μετά την άφηξή τους. Ακούσαμε και τους τρόπους ε, με τους οποίους ε, ε, είναι πιο ευάλωτες οι γυναίκες και μάλιστα δυσανάλογα και επίσης από τις έρευνες γνωρίζουμε ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι σχετικά χαμηλά στις προτεραιότητες. Το να βρουν στέγη, να επανενωθούν με τις οικογένειές τους είναι οι πρώτε τους προτεραιότητες και γνωρίζουμε ότι ένα καλό περιβάλλον επανεγκατάστασης, απασχόληση, οικογενειακή επανένεση, προστασία κατά των διακρίσεων και να μην υπάρχει Όλα αυτά δημιουργούν σε καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία. Αυτό αποδεικνύεται και μπορούμε να αποδείξουμε και ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα συμβεί ε, με ε, πολλαπλές εργασίες ή με ενιαίες θηρίδες όπου ε, θα συναντούν οι επαγγελματίες στην υπηρεσία στον τομέα της υγείας τις γυναίκες πρόσφυγες μαζί, όχι να έρχονται οι γυναίκες πρόσφυγες να συναντήσουν τον καθένα ξεχωριστά. Υπάρχει το θέμα της διερμηνίας μεν, υπάρχει μεταφορά, ε, μετάφραση και συμβουλές και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται σε μια ατμόσφαιρα που θα παρακινεί περισσότερο προς την αποδοχή και όχι ε, ε, στο στίγμα. Ε, θα μιλήσω και λίγο για τις ανάγκες. Εγώ θα προτείνω κάποια πράγματα, παρόλο που δεν μου ζητήσετε. Προτείνω καταρχάς να μην υπάρχουν νομικοί περιορισμοί για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Να υπάρχει κατάλληλη κάλυψη για εγγύους και για παιδιά, ε, ανεξάρτητα από το καθεστώς που τους δίνει τους πρόσφυγες ή μετανάστες, ε, ε βελτίωση στην ε, διερμηνία, τεκμηρίωση για τους ασθενείς, ώστε να μην πρέπει συνεχώς να περιγράφουν την κατάστασή τους ε, και εκεί φυσικά έρχεται και το ψυχολογικό σκέλος που έρχεται να συσσωρευτεί στην τραυματική κατάσταση που βιώνουν και φυσικά ε, προστασία για πιο ευάλωτες ομάδες με τρόπους ε, που θα τους υποστηρίξουν ώστε να αντέξουν και θα αποφύγουν το στίγμα. Οι γυναίκες αυτές αντέχουν με πάρα πολλούς τρόπους που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε με τα συνήθη τεστ υγείας. Επίση, να υπάρχουν κάποια μοντέλα υγειονομική περίθαλψη, ε, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη ότι ε, πλέον είναι το σύνηθε ε, η κινητικότητα. Η κρίση των προσφύγων υπονοεί ότι κάπως θα, θα σταματήσει και όντω κάποια πράγματα θα σταματήσουν, η πίεση του πολέμου. Αλλά η κινητικότητα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι χαρακτηριστικό του κόσμου μας και τη κοινωνία μα για πολύ μεγάλο διάστημα από εδώ και πέρα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you so much, Professor Ευχαριστώ. Καθηγητά Μπράντμπι. Και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Κιάρα Μοντάλτο, την τρίτη δική μας. Εκπροσωπεί μια πολύ σημαντική μη κυβερνητική οργάνωση. Και θα δώσει μαρτυρία, πιστεύω, πολύτιμη για τη δουλειά Μπορείτε να λάβετε το λόγο κυρία Μοντάλτο. Ναι, ευχαριστώ. Έχω κάποιες ε, διαφάνειες προβλέψεις, αλλά μάλλον κάποιο τεχνικό πρόβλημα θα, μας επιτρέψει να τις δείξουμε. Να ξεκινήσω ίσως πρώτα. Θα ξεκινήσω με τη μικρή μου σύντομη αυτή ομιλία. Η ειδική δεν ξέρω αν πρέπει να με πει κανείς Περισσότερο μάρτυρας είμαι παρά εμπειρογνώμων. τις μάρτυρες γιατί βρίσκομαι εκεί στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σερβία δουλεύω. Πρόσφατα στη Μυτιλίνη στην Ελλάδα. Και θα προσπαθήσω σήμερα να σας περιγράψω αυτά που καθημερινά βλέπω και να μετατραπώ στη φωνή των ανθρώπων αυτών που συναντώ κάθε μέρα. Για να σας δώσω μια σύντομη ιδέα της δράσης μας και να περάσω στην επόμενη διαφάνεια. Το 2015 στην Ελλάδα και τη Σερβία είδαμε 100.000 περίπου άτομα ως γιατροί. Θα δείτε εδώ λοιπόν τι τύπο ασθενών ε, δεχθήκαμε στο δρόμο των Βαλκανίων και τη Σικελία. 20% όπως βλέπετε των ε, ανθρώπων που βλέπουμε είναι γυναίκες, 1% εξ αυτών έγκυοι. Επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο στους α, μη συνοδευόμενους ανηλίκους είχαμε 3% κορίτσια που δεν το είχαμε δει νωρίτερα. Πολύ μεγάλο ποσοστό λοιπόν, ανησυχητικό ποσοστό και μιλώ για πραγματικούς μη συνοδευόμενου νέους, όχι αυτού που θα έλεγε κανεί ανηλίκους είναι, ακόμα, είναι 17-18 ετών τυπικά, είναι ανήλικοι κτλ. Μιλώ για πολύ μικρές ηλικίε. Και αυτές είναι οι δικέ μας οι, τα δικά μας τα ραντεβού τα ιατρικά. Ε, φυσικά δεν μπορώ να πω ότι ισχύει το ίδιο παντού. Είναι η απεικόνηση η δική μου αυτό που σας παρουσιάζω και στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό προσπαθούμε να προσφέρουμε είναι η ιατρική ε, φροντίδα αφού είμαστε βέβαια ιατρική οργάνωση ιατρών, ιατροί χωρίς σύνορα και ή δυνατόν ε, να καθοδηγήσουμε προς νοσοκομιακή περίθαλψη αν χρειάζεται. Ωστόσο αυτή η ιατρική περίθαλψη δεν είναι μόνο να δώσω ένα χάπι για μένα. Είναι κάτι το πολύ περισσότερο, κάτι το πολύ διαφορετικό, όπως είπε και η συνάδελφος νωρίτερα, η υποστήριξη, η παρακολούθηση, η στήριξη από διαμεσολαβητή αυτού του τύπου που σε τελευταία ανάλυση παίζει και το ρόλο του ψυχοθεραπευτή, εκείνου ο οποίος θα παίζει το ρόλο του ε, συνδετικού κρίκου γιατί θα μιλάει τη γλώσσα του, του διερμηνέα δηλαδή, είναι πολλές φορές σωτήρια και απαραίτητη. Όταν χρειάζεται στέλνουμε τους ασθενείς μας στα νοσοκομεία, αλλά θα σας το πω και εκτενέστερα πιο μετά, αρνούνται οι περισσότεροι την νοσηλεία, το επεσήμανε και η συνάδελφος πριν, γιατί η νομική τους κατάσταση είναι το κύριο εμπόδιο που έχουν να αντιμετωπίσουν και δεν τους επιτρέπει καν να πάνε να ζητήσουν βοήθεια ή ιατρική περίθαλψη. Ξέρουμε πολύ καλά από τι τραυματικές εμπειρίες έχουν περάσει οι άνθρωποι αυτοί. Είναι πολύ σημαντικό η ιατρικη περιθαλψη ξερουμε πολυ καλα απο τι τραυματικες εμπειριες εχουν παρασει οι ανθρωποι αυτοι ειναι πολυ σημαντικο η ομαδα μας να τους προσφέρει όχι μόνο ιατρικό προσωπικό γιατρό νοσοκόμα αλλά και την ε, ψυχολογική υποστήριξη, την ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζονται. Αυτό δεν είναι εύκολο βέβαια. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι περνάνε πολύ γρήγορα και δεν έχουν χρόνο να μας αφιερώσουν γιατί οι προτεραιότητες είναι άλλοι. Ωστόσο προσπαθούμε όσο μπορούμε να αναπτύξουμε μια ψυχολογική μια υπηρεσία ψυχολογικών πρώτων βοηθειών, που δεν είναι σωστό όρο, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ψυχολογική στήριξη, αλλά μια δραστηριότητα που θα επιτρέψει απλώ το μετριασμό του οξέου τραύματο τη στιγμή. Δεν λύνουμε τα ψυχολογικά προβλήματα των ανθρώπων αυτών, δεν του βοηθούμε να αντιμετωπίσουν τα ψυχολογικά του τραύματα. Ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν στι χώρε προορισμού, μακροπρόθεσμα. Αλλά εμεί πάνω στον δρόμο αυτόν, ε, ε, στην πορεία του, προσπαθούμε κάπω να του ανακουφίσουμε. Την επόμενη διαφάνεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ανάγκε των ανθρώπων δεν έχουν μόνο ιατρικό χαρακτήρα και όταν οι ιατρικέ ανάγκε ε, είναι και για αυτού ακόμη μπορεί να είναι σημαντικέ, σημαντικά προβλήματα υγεία, πάλι δεν είναι προτεραιότητα γιατί χρειάζονται πρώτα απ' όλα ένα κατάλημα, ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα, και μια, ε, ένα, ιατρικό, ένα νομικό καθεστώ, αναγνωρισμένο καθεστώ. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να οργανώσουμε, να προσφέρουμε ένα, κατα... ένα κατάλημα και με θέρμανση που δεν ήταν δεδομένο ούτε στην Σερβία αλλά ούτε καν στην Ελλάδα. Είχαμε και υποθερμίες, είχαμε και κρυοπαγήματα. Ε, προσπαθούμε να δώσουμε επίσης και ε, αντικείμενα τα οποία δεν είναι μόνο τρόφιμα όπως ε, κουβέρτες, ρουχ, ρουχισμό, τρόπο μεταφοράς ακόμη από το ένα σημείο στο άλλο. Όσο μπορούμε δηλαδή οργανωμένο και πλήρες πακέτο υπηρεσίας και αυτό σε συνεργασία και συντονισμό με άλλους παράγοντες που δραστηριοποιούνται. Δεν είμαστε ούτε ικανοί, ε, ούτε καν έχουμε τη δυνατότητα και την εντολή να το πράξουμε αυτό συνολικά. Και έχουμε αναλάβει ακόμη και δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, τώρα όλο και περισσότερο στο Αιγαίο. Όπως ξέρετε όλο συνεχίζονται οι νεκροί και στο Αιγαίο είναι για μας ακόμα μεγαλύτερος ε, ο, ο κλονισμός που ε, ε, ζούμε γιατί η Τουρκία, τα, η, η στεριά η τουρκική είναι σε ορατή απόσταση. Δεν υπάρχει όμως τρόπος νόμιμος και ασφαλής να περάσουν οι άνθρωποι αυτοί. Και παρόλα αυτά παίρνουν πάνω από χίλια άνθρωποι κάθε μέρα παίρνουν το δρόμο αυτόν με τα ελαφρά πλοιάρια για να φτάσουν στις ελληνικές ακτές. Φυσικά ό,τι και να κάνουμε θα παραμείνει στον αέρα εάν δεν ανοίξουμε το θέμα, αν δεν υποστηρίξουμε, αν δεν μιλήσουμε ανοιχτά. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα για να αλλάξουν οι νοοτροπίες και οι στάσεις απέναντι στην προσφυγική κρίση. Ιδιαίτερα εστιαζόμαστε στις γυναίκες γιατί είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα με τη σημερινή μας τοποθέτηση ε, βλέπετε εδώ ότι από τις γυναίκες έχουμε κυρίως ε, αναπνευστικά προβλήματα, γαστροεντερικά προβλήματα. Ένα 10 περίπου της ε, έχει φέρει τραύματα και πληγές λόγω βίας, είτε στη χώρα προελεύσεως είτε στη χώρα διελεύσεως και μάλιστα όχι μόνο πριν να φτάσουν σε ευρωπαϊκά εδάφη αλλά και μέσα στην Ευρώπη. Αυτό που είναι πραγματικά τρομακτικό και εντυπωσιακό είναι ότι το περισσότερο από το μισό από τα ε, επεισόδια αυτά βίας βλέπουμε να ασκείται από θεσμικούς φορεί. θα το πω έτσι, εντυπωσιακό ποσοστό. Επίσης έχουμε και χρόνιες ασθένειε, γιατί ανεβαίνει συνέχεια η ηλικία αυτών των ανθρώπων και των γυναικών ιδιαίτερως και έτσι αντιμετωπίζουμε ε, ασθένειες που δεν είχαμε πριν ε, το 2004. Τώρα βλέπουμε και πολλούς ασθένειες με διαβήτη, με καρδιαγκιακές παθήσεις, με πνευμονικές παθήσεις, χρόνιες. Προσπαθούμε να δώσουμε στο δυνατόν καλύτερη ε, αγωγή έτσι ώστε να τους ετοιμάσουμε και όταν φτάσουν στην χώρα προορισμού να έχουν την κατάλληλη περίθαλψη. Βέβαια τους δίνουμε και ιατρικό πιστοποιητικό εφόσον αυτό ελπίζουμε μπορεί να τους φανεί χρήσιμο για να έχουν ταχύτερη και καλύτερη αντιμετώπιση, αν και αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο, οι χώρες προορισμού πολλές φορές δεν είναι οι γη της επαγγελίας που περιμένουν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς ε, σε αυτή την πορεία να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε. Και επίσης ε, πέραν αυτού έχουμε πολλά προβλήματα που δεν θέλω να πω ότι είναι ε, είναι ψυχολογικά προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, όπως και να τα πούμε. Έχουν περάσει πολλές τραυματικές εμπειρίες. Είναι πάρα πολύ ε, φυσιολογικό να δει κανείς υψηλά ποσοστά εκδηλώσεων συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης, μετατραυματικής κατάθλιψης, ε, δυσκολία προσαρμογής ή πολύ έντονες αντιδράσεις. Όλα αυτά που ξέρουμε ότι θα χρειαστούν και περαιτέρω αντιμετώπιση. Τελειώνω σχεδόν από τις γυναίκες αυτές. 10% έρχονται έγκυοι ή λεχόνες. Έχουν γεννήσει στο δρόμο. Κοιτάμε φυσικά να δούμε, να ελέγξουμε τα παιδιά τους ότι είναι καλά στην υγεία τους. Πολλές φορές όμως και είναι τρομακτικό αυτό. Ακόμα και πολλοί άρρωστες να είναι αρνούνται την, την ε, ε, νοσηλεία. Πριν από δύο μήνες ήμουνα στην ειδωμένη μεταξύ Ελλάδα και Σερβίας, λέει η ομιλήτρια. Έφτασε μέσα σε μια πολύ κρύα νύχτα του χειμώνα μια γυναίκα με επτά μήνες εγκυμοσύνη, με, βαρύτατη, ε, με βαρύτατο ύκτερο, κίτρινη σαν το λεμόνι, δεν δέχθηκε να πάει στο νοσοκομείο όπως εμείς θέλαμε, συνέχισε το δρόμο της και ε, ε, έλεγε δεν μπορώ να ξεφύγω από την ομάδα μου, δεν μπορώ να χάσω την ομάδα μου, πρέπει να προχωρήσω μαζί τους πριν κλείσουν τα σύνορα, γιατί ακόμα ήταν ανοιχτά κάπως τα σύνορα εκείνη την εποχή. Και ακόμα σκέφτομαι τι της συνέβη, τι, ποια ήταν η μοίρα της εκείνης και του παιδιού της. Μία από τόσους πρόσφυγες άλλα. Όπως είπα, πολλοί, είναι, πολλές είναι αυτές οι οποίες ακόμη και σε πολύ κακές κλινικά καταστάσεις αρνούνται την οσυλία και την περίθαλψη. Για να ολοκληρώσω. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται πράγματι βοήθεια. Όχι με βάση την εθνικότητα, όπω δυστυχώ βλέπουμε να συμβαίνει τώρα, αλλά με βάση τι ατομικέ του ανάγκε να εξασφαλίσουν προστασία. Γιατί έχουν παρελθόν ευάλωτων καταστάσεων, τραυματικές εμπειρίες που ανέφερα νωρίτερα. Έχουν όλους τους επιβαρυντικούς παράγοντες, στο ε, δρόμο της μετανάστευσης, την απουσία περίθαλψης, καταλήματος κατάλληλου, τροφής, αξιοπρέπειας ακόμη, όλα αυτά τα οποία συζητούμε. Και κλείνοντας, θα ήθελα να φέρω ένα άλλο παράδειγμα, με το οποίο βρέθηκα τη μέτωπη πάλι στην Εδωμένη, ένα παιδί, ένα κοριτσάκι, 7 ετών, από το Ιράν, μέσα σε όλο αυτό το χάος της Εδωμένης, ήταν το κοριτσάκι αυτό, η μαμά της μου έδειξε το ιατρικό πιστοποιητικό, είχε βαρύτατη καρδιακή ανεπάρκεια, χρειαζόταν μεταμόσχευση καρδιάς, και μαζί της όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά, εγώ είδα το παιδί, είδα τα πιστοποιητικά και ζήτησα από όλες τις παρούσες υπηρεσίες να της δώσουν την προστασία και η απάντηση όχι γιατί είναι αυτό το Ιράν. Αυτό το παιδί άλλη επιλογή δεν είχε παρά μόνο να βάλει τη ζωή του στα χέρια των λαθροδιακινητών, μπα και φτάσει σε κάποια χώρα που θα μπορούσε κάποιο γιατρό να τη σώσει τη ζωή. Απαράδεκτο αυτό για μα. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται προστασία, όχι γιατί έχουν κάποια πινακίδα στο, στο μέτωπο που λέει με πρόσφυγα, αλλά γιατί βρίσκονται σε κατάσταση ε, επικίνδυνη, γιατί έχουν εκτεθεί σε κινδύνους, γιατί είναι ευάλωτοι. Και κλείνοντας με τελευταία σελίδα της παρουσίασής μου, θέλω να μιλήσω για το hashtag ασφαλής διέλευση, safe passage. Αυτό δεν σημαίνει βάλτε περισσότερα ε, σκάφη στην, ε, στο Αιγαίο, αλλά εξασφαλίστε νόμιμους τρόπους διέλευσης για τους ανθρώπους αυτούς, γιατί διακινδυνεύουν τη ζωή τους αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Δεν θα σταματούμε ποτέ να το επαναλαμβάνουμε, αλλά πρέπει να σας πω ότι τώρα αισθανόμαστε μεγάλη δυσφορία και απόγνωση γιατί χρόνια τώρα το λέμε, δεν αλλάζει τίποτα ή μάλλον όχι, τα πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο. Είναι τρομακτικό το ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που φέρουν στην ειδωμένη. Κάθε μέρα φτάνουν χιλιάδες πρόσφυγες. 13.000 είναι σήμερα. Χωρίς κατάλημα, χωρίς καταφύγιο, μέσα στη βροχή και το κρύο. Σας ευχαριστούμε κυρία Μοντάλντο. Τώρα δίνω την Προεδρία στην Συμπρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την προλαλήσασα για την ε, εισαγωγή. Τώρα έχετε εσείς κυρίες μου και κύριοι το λόγο όσοι ζήτησαν. Κυρία Ματάη από την ε, Ουγγαρία πρώτα έχει στήσει το λόγο, θα δώσουμε στη συνέχεια και στους υπόλοιπους ενδιαφερμένους. Σας παρακαλώ όμως να μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά για να δώσουμε το λόγο σε όσο το δυνατόν περισσότερες και περισσότερους ομιλητές. Η κυρία Μάτραη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Γιατί οι προσεγγίσεις του παρελθόντος και οι πολιτικές του παρελθόντος δεν λειτουργούν πια σήμερα. Έχουμε πολύ μεγαλύτερες υγειονομικές ε, προκλήσεις. Στην Ουγγαρία το 2015 είχαμε άφεξη πάνω από 150.000 προσφύγων έτων τον άσυλο. Ένα, ένα αριθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης, ε, μέσα σε μια εβδομάδα η πλειοψηφία τους ε, υπέβαλε αιτήσεις, υπέβαλε αιτήσεις ασύλου στις αρμόδιες αρχές και η Ουγγρική κυβέρνηση έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και από υγειονομική άποψη και οι πιο ευάλωτοι, οι γυναίκες κυρίως και οι ανήλικοι, είναι αυτοί που χρήζουν άμεσες βοήθειες. λήφθησαν υπόψη. Βέβαια υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές και ιδεολογικές και πολιτισμικές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πολλές γυναίκες αρνούνται η υγειονομική περίθαλψη ή έστω και επίσκεψη στο γιατρό όταν αυτός είναι άντρας. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ευαισθησίες. Το 20% των ετουσών άσυλο έχουν ήδη λάβει μια απάντηση φέτος. και όσοι έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου ήδη δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη και επίσκεψη σε ένα παθολόγο. Οι υπόλοιποι μόνο όταν υπάρχει κάτι επίγον. Δικαιούνται μόνο σε επίγον περιστατικό κάποια υγειονομική περίθαλψη. Πάντως ε, υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και μάλιστα με ίδιους όρους με τους Ούγγρους πολίτες. 200.000 ευρώ μας κόστισε αυτή η πρόσβαση πέρυσι. Οι περισσότεροι είναι νέοι. Ένα μικρό ποσοστό έχει σοβαρέ ασθένειε και κάποιοι έχουν και αναπηρίες. Αλλά διαπιστώσαμε ότι οι πλέον ευάλωτες είναι οι γυναίκες. Η πρόεδρος διακόπτη γιατί έχει ξεπεράσει το δίλεπτο. Πάντως δεν έχουμε πολλές πληροφορίες ακόμη. Θα πρέπει να, να ενημερώνονται καλύτερα οι πρόσφυγες και μετανάστες για τις δυνατότητες που έχουν να αποταθούν σε γιατρό ή να τύχουν υγειονομικής περίθαλψης. Πάντως σήμερα ένα, ένα τρίτο των μεταναστών και προσφύγων είναι γυναίκες, το 50% είναι έγκυες. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε πολύ περισσότερα στοιχεία και κυρίως να δούμε ποιες είναι οι αρνητικέ συνέπειες αυτής της μετακίνησης για τις γυναίκες και να τις αντιμετωπίσουμε. Σας ε, ευχαριστώ. Σας παρακαλώ όμως και να σεβαστείτε το χρόνο για να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις από εσά και να λάβουμε συγκεκριμένες απαντήσεις από τις ομιλητριές μας. Είναι νομίζω σωστό να διαχειριστούμε το χρόνο μας έτσι ώστε να μιλήσουν και οι άλλοι. Η κυρία Ντοάν έχει το λόγο. Öncelikle Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τι ευχαριστίε μου και την ευγνωμοσύνη μου για τη δυνατότητα που μα προσφέρεται να είμαστε σε μια τέτοια σε μια πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συζητάει τόσο σημαντικά θέματα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω χαιρετισμό για την ε, Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας. Έχουμε από το 2011 πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών οι οποίες έφυγαν από τη Συρία και έχουν εγκαταστεί πρόσφυγες ε, και στην Τουρκία και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου και αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Η Τουρκία είναι μία από τις χώρες οι οποίες τις υποδέχεται σε πολύ μεγάλους αριθμούς και αντιμετωπίζει και εκείνη από την πλευρά της πολλές δυσκολίες. Θα ήθελα εδώ να ζητήσουμε μάλιστα να μιλήσουμε και για την ε, θετική προτίμηση. Μαζί με τους ε, Σύρους αλλά και τους Ιρακινούς οι, οι πρόσφυγες που δέχεται η Συρία είναι πολύ άριθμοι πάνω από 150.000 Σύριοι πρόσφυγες αλλά και Ιρακινοί βρίσκονται στις πόλεις μας. Η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες μιλάει για 19 εκατομμύρια πρόσφυγες ανά τον κόσμο, εκ των οποίων 3, 3 εκατομμύρια συνολικά βρίσκονται στην ε, Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η Τουρκία έχει δαπανίσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών για τους πρόσφυγες που υποδέχεται. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι γυναίκες, τα παιδιά χαρακτηρίζονται από όλους τους ειδικού ως ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες ε, μεταξύ των ομάδων των προσφύγων. Οι γυναίκες ε, και λόγω του ρόλου που έχουν στην οικογένεια αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερες πιέσεις και δυσκολίες. είναι θύματα των πολέμων, των συγκρούσεων, πέφτουν θύματα ε, της σεξουαλικής ε, βίας και των βιασμών. Πολλές φορές έχουν χάσει τα πάντα οι γυναίκες αυτές και αναζητούν νέες ευκαιρίες ε, σε μια νέα χώρα, πέφτουν όμως θύματα της εκμετάλλευσης και των διακινητών μια από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές που έχουμε αναπτύξει εμείς στην Τουρκία και νομίζω το αποδέχεται ολόκληρος ο κόσμος είναι η πολιτική σχετική με την ετροφαρμακευτική περίθαλψη και στο επίπεδο αυτό έχουμε εξασφαλίσει πολύ, σημαντικές, πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Θα ήθελα να σας δώσω λοιπόν τα πορίσματα ενός ε, σεμιναρίου που κάναμε για το θέμα αυτό της φαρμακευτικής περίθαψης για τις γυναίκες ε, πρόσφυγες στην Τουρκία. Ανεξαρτήτως του καθεστώτος που έχουν λάβει, πρόκειται για πρόσφυγες ή για μετανάστες λοιπόν. Όποιες γυναίκες είχαν ανάγκη από υποστήριξη και προστασία στην Τουρκία, είχαν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία υγείας ιατροφαρμακευτική που έχει και η υπήκος. Ε, η γυναίκα υπήκοσης Τουρκίας. Και αν θέλετε μπορώ να σας και πιο πολλές λεπτομέρειες. Η πρόεδρος ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την ενημέρωση από την Τουρκία και καλό την επόμενη ομιλήτρια. Μαρία Πάου Ελληνιγέννη και ελπίζω να έχω προφέρει σωστά το όνομά σας. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές ε, αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης και τους ευχαριστούμε για την πρόσκληση οι γυναίκες και τα κορίτσια που ζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα της αναπαραγωγικής τους υγείας θα γίνουν σεβαστά. Παρ' όλα αυτά, μερικές ευρωπαϊκές χώρες ε, δεν σέβονται τα γυναικεία δικαιώματα ή τα αναπαραγωγικά δικαιώματα ή τα περιορίζουν. Η Λιθουανία δεν έχει ακόμη... Ε, ε, ούτε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ούτε νομοθεσία για την ε, ε, ιατρικώς υποβοηθούμενη γονιμοποίηση. Οπότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα θέματα του φύλου και ε, τα θέματα αυτά τα, ε, της υγείας σε μια Ευρώπη που παρουσιάζει έξαρση, η μυσαλλοδοξία, η τάση κατά των μεταναστών και ξενοφοβία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ντορίν Μασέη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση. Έχω κάποια σχόλια και μερικές ερωτήσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες είναι το θεμέλιο πολλών οικογενειών και η αντιμετώπιση δική τους θα έχει, θα έχει αντανάκλαση και στα παιδιά τους και Πολλές φορές είναι θύματα βίας και σεξουαλικής, θύματα υποσυτισμού, ε, ψυχολογικού άγχους. Τα παιδιά γίνονται μάρτυρες αυτών των ε, δεινών και ε, τραυματίζονται από τα δεινά των μητέρων τους. Αυτό πραγματικά είναι κρίμα, γιατί γνωρίζουμε από τις έρευνες πόσο περίπλοκες είναι οι ανάγκες των γυναικών. Μερικές φορές έχουν και ψυχολογικά προβλήματα. Και το θέμα της ένταξης στις νέες κοινωνίες ε, προϋποθέτει και μία στήριξη και σε θέματα ε, εκμάθησης γλωσσών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ ψηλότερη η ανεργία των γυναικών και φυσικά όλες αυτές οι αρνητικές συνέπειες ε, θα επηρεάσουν τα παιδιά. Η Επιτροπή Ιστορικών Υποθέσεων της Βουλής των Λόρδων ξεκίνησε μία έρευνα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Τι είστε όμως ανήλικος. Μπορεί να είναι ένα αγόρι, ένα κορίτσι 17 ετών οι περισσότεροι ενηλικοί είναι συνήθως ε, παιδιά προς κοντά στην ενηλικίωση με τα γνωστά εφηβικά προβλήματα. Θα πρέπει να ακούσουμε τη φωνή και αυτών των εφήβων, αυτών των ανηλίκων. Και αν κανείς ε, έχει τέτοια στοιχεία, πολύ θα θέλαμε να τα ακούσουμε. Νομίζω θίξατε ένα πολύ, πολύ σημαντικό τομέα. Κυρία Αλίνα Τελτιάλα, από την Αλβανία. Σα Σας ευχαριστώ. Η σημερινή κατάσταση δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις για ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ξαναρχίζω. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, επαναλαμβάνω λοιπόν, η σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη δημιουργεί προκλήσεις για όλες τις χώρες. Η Αλβανία έχει σήμερα 60.000 πρόσφυγες, 20% αυτών είναι γυναίκες. Το 2015 ήταν το έτος των προσφύγων στην Αλβανία. Η αλβανική κυβέρνηση φαίνεται να θελοτυφλεί, αρνείται το πρόβλημα και θεωρεί ότι είναι απλώς πρόβλημα συνοριακό μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας και η Αλβανία υποφέρει από την σύραξη στη Συρία. Γιατί και η Αλβανία έχει προβλήματα. Γιατί και στη χώρα μου οι γυναίκες υποφέρουν. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα των προσφύγων οφείλεται μόνο στην κακή διακυβέρνηση, στην έλλειψη ευκαιριών ή στην έλλειψη απασχόλησης. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο ε, ευαίσθητες, ε, φροντίζουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους και υποφέρουν πολύ περισσότερο όταν ξεκινούν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι αναζητώντας προστασία και καταφύγιο σε μια άλλη χώρα. Και οι υπηρεσίες υγεία έχουν κέρια σημασία, γιατί οι γυναίκες πρόσφυγες και τα κορίτσια πρόσφυγες είναι πιο ευάλωτες στους κινδύνους και υποφέρουν ε, τα πάνδυνα σε αυτό το ταξίδι προς την Ευρώπη. Πολλές φορές ε, έχουν τραυματικές εμπειρίες, ε, ψυχολογικά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να άρουμε τα εμπόδια και τη γραφειοκρατία και να προσφέρουμε υγειονομική περίθαλψη έγκαιρα στις γυναίκες και τα κορίτσια που τη χρειάζονται. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διάσταση του φύλου και γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβουμε υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών που υποφέρουν περισσότερο μέσα σε αυτά τα προσφυγικά και μεταναστευτικά κινήματα. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να καταργηθεί η γραφειοκρατία και να εξασφαλίζεται πολύ πιο άμεση πρόσβαση και υποδοχή των γυναικών στις χώρες προορισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως για την συνδρομή που έχουν προσφέρει τους Αλβανούς μετανάστες και πρόσφυγες και τον άσυλο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις για όλες τις χώρες και για την Αλβανία και θα πρέπει πολλά να αλλάξουν ώστε και οι Αλβανοί να αισθάνονται καλοδεχούμενοι. Η κυρία Γκόρδανα Σόπολ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Είμαι από την Κροατία. Είναι μία από τις χώρες του Βαλκανικού διαδρόμου ή της Βαλκανικού οδού, αυτού του τεράστιου προσφυγικού κύματος. Από τα, από τα μέσα του προηγούμενου έτους πέρασαν από την Κροατία περίπου 550.000 πρόσφυγες και μετα, μετανάστες. Ε, περίπου 20 από αυτούς είναι γυναίκες ενήλικες. Τώρα για τους ανήλικους, για τα παιδιά, έχουμε κορίτσια, το 40% αυτό είναι περίπου κορίτσια. Αυτό που αντιμετώπισε η πατρίδα μου η Κροατία, καταρχήν νομίζω ότι η χώρα μου ήταν υπόδειγμα σωστής περίθαλψης αυτών των ε, τεράστιων κυμάτων των προσφύγων. Ε, μέχρι στιγμής μόνο 24 ε, ζήτησαν άσυλο στην ε, Κροατία, 22 από αυτούς είναι άνδρες και δύο μόνο γυναίκες ζήτησαν άσυλο στην Κροατία. Εμείς φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε στέγη, κατάλημα και υγειονομική περίθαψη στους πρόσφυγες αυτούς. Μερικές φορές όμως, μερικοί αρνήθηκαν ακόμη και την εισαγωγή ή την ασυλία γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε για αυτούς απομάκρυνση είτε από την οικογένεια ή από την ομάδα με την οποία έφτασαν στην Κροατία και γι' αυτό απέρριψαν, αρνήθηκαν την οσυλία. Είχαμε και τέτοια παραδείγματα. Δεν ήθελαν με μια πιθανή εισαγωγή στο νοσοκομείο να χάσουν χρόνο και να επιβραδύνουν την άφηξή τους στη χώρα προορισμού. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μεριμνήσουμε για τους πρόσφυγες αυτούς και Όπως είπαμε, κάποια στιγμή θα φτάσουν στη χώρα προορισμού. Τότε τα, προβλήματα υγείας και τα ψυχολογικά προβλήματα δεν θα τα έχουν ξεπεράσει. Τότε είναι που θα φανούν περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον να προσανατολιστούμε προς την επίλυση και αυτού του πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη έκκληση, πραγματική δουλειά να ξεκινήσει τελικά. Η κυρία Κέντζη έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, ε. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για αυτή την τόσο σημαντική ημέρα που έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή. Θα πάρω το λόγο αργότερα και στην Ολομέλεια για να παρουσιάσω την έκθεση πρωτοβουλίας ε, για την ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση και το άθυλο, στην οποία φυσικά περιλαμβάνεται και μια ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τα προβλήματα των γυναικών. Θα ήθελα εδώ να επιστήσω την προσοχή σας ε, στο θέμα της υγειονομικής περίθαλψης. Είμαι ιατρός, ε, οφθαλμίατρος, Επομένως, ε, στη ζωή μου έχω ασκήσει και τη δραστηριότητα που υπενθύμησαν και οι συνάδελφοι που αφορά τη βοήθεια προς τις γυναίκες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη σημαντική πορεία των γυναικών και κυρίως την υγεία τους. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και κυρίως την ψυχική τους υγεία υγεία. Πολλές από αυτές τις γυναίκες φτάνουν εδώ ε, μετά από βιασμό, ε, μετά από ανθρώπους που ε, ε, τις είχαν κακοποιήσει. Γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τις γυναίκες τις εκμεταλλεύονται σε όλες τις συνθήκες. Αλλά σε αυτή την πορεία φυγής από τη χώρα καταγωγής τους ε, χρησιμοποιούνται και ως όπλο ανταλλαγής που χρησιμοποιούν οι διακινητές. φτάνουν, χρειάζονται πρώτες βοήθειες στην πραγματικότητα. Ε, πρέπει να ολοκληρώσω βλέπω. Χρειάζεται ε, να τους παρασχεθεί άμεση βοήθεια όσον αφορά την ε, ψυχική τους υγεία και εμείς πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα θέματα αυτά. Και όχι μόνο αυτά. Τα τα παιδιά συγγνώμη, που γεννούνται από βιασμένε γυναίκε είναι ένα εντελώ ξεχωριστό κεφάλαιο, διότι πολλά από αυτά τα παιδιά ε, γεννιούνται από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Επομένω, η κοινωνία μα πρέπει να αναρωτηθεί λίγο για το μέλλον αυτών των παιδιών. Και η διάσκεψη εδώ θα πρέπει να λάβει υπόψη τη και τι γυναίκε, αλλά και τα παιδιά τα οποία γεννούν αυτέ οι γυναίκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε, άμα προσέχουμε το χρόνο, γιατί έχουμε μόνο πέντε λεπτά ακόμα μέχρι να ξαναμπούν οι υπόλοιπε προσκεκλημένε μα και οι προσκεκλημένοι στην αίθουσα. Τώρα θα πρέπει να περιοριστούμε στον ένα. Στο ένα λεπτό η κυρία Ολρίκε Χίλε η επόμενη. Ναι, ευχαριστώ και εγώ για την διάσκεψη για τη σημαντική αυτή εκθέση. Θα ήθελα να δείξω τρία σημεία. Καταρχάς, συγκεκριμένα, για την επανεγκατάσταση. Τι θέση έχετε διότι το πρόγραμμα επανεκατάστασης με το Ινήπατη Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες επιτρέπει να φτάσουν ταχύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια οι πρόσφυγες στο υλικό τους προορισμό και να μην περάσουν αυτόν τον αποτρόπαιο δρόμο της φυγής. Το άλλο σημαντικό για μένα είναι η επανένωση των οικογενειών, αν υπάρχουν δυνατότητες. Για γυναίκες βέβαια και για παιδιά πάνω απ' όλα, πρέπει να καταφέρουν να φτάνουν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια στην Ευρώπη. Εμείς στη Γερμανία ξέρουμε ότι πολλές φορές έρχονται πρώτα οι άντρες και έχουμε μεγάλο δημόσιο διάλογο στη Γερμανία σχετικό με την επανένωση των οικογενειών. Και τελευταίο, πολύ σύντομα, τα αίτια της φυγής, τα αίτια της προσφυγιάς. Είναι φρικτός ο πόλεμος στη Συρία και στο γυναικείο κίνημα πάντοτε ε, αγωνιζόμασταν και για τη, υπέρ της ειρήνης, όχι μόνο σήμερα, αλλά πάντα γενικότερα. Προσπαθούσαμε να κάνουμε περισσότερα ως μια ευρωπαϊκή κοινότητα αξιών για την ανθρωπιά και για την ειρήνη. Θέλαμε να υψώνουμε πάντα τη φωνή μας και να μιλούμε υπέρ της ειρήνης. Ιδάλλως πάντα θα έχουμε αφόρητες καταστάσεις προσφυγιάς. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Νικόλα. Μαυρό Νικόλα, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι από την Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή δεν είναι χώρα προορισμού για τους πρόσφυγες λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Όμως ξέρουμε πολύ καλά εμείς στην Κύπρο τι σημαίνει προσφυγιά και πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, η πρώτη ανάγκη αυτών των ανθρώπων που φεύγουν από την πατρίδα τους για να σωθούν ε, δεν είναι ασφαλώς για να μεταναστεύσουν ούτε για να ζήσουν καλύτερα αλλά είναι να νιώσουν ασφάλεια και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι πάντα τα μεγαλύτερα θύματα. Χάνουν την ταυτότητά τους, χάνουν την αξιοπρέπεια τους και είναι πολύ σημαντικό το πώς νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος περιμένει στην ουρά για μια κουβέρτα, για ένα κομμάτι ψωμί, για να ζήσει και να επιβιώσει μαζί με τα παιδιά του. Ε, άρα θεωρώ ότι η κακοποίηση αυτών των ανθρώπων είναι και ψυχολογική, είναι και σεξουαλική, είναι και σωματική. Άρα πέρα από την υγεία όπως την αντιλαμβανόμαστε να τους ε, ηρεμήσουμε τις πληγές τους θα πρέπει να δούμε και τη ψυχική υγεία αυτών των ανθρώπων γιατί εκείνος ο οποίος είναι πρόσφυγας δεν ξεχνά ποτέ και να πω ότι εμείς στην Κύπρο και πρέπει θέλω να το ρωτήσω αυτό υπάρχουν ε, γυναίκες οι οποίες έμειναν έγκυες ασφαλώς από σεξουαλική κακοποίηση τι γίνεται με αυτές τις γυναίκες. Έχουν την ευκαιρία και το περιθώριο εάν θέλουν να κάνουν έκτρωση ή πρέπει να, να μείνουν έγκυες να γεννήσουν αυτά τα παιδιά με όλα αυτά τα επακόλουθα που όλες μας γνωρίζουμε. Εμείς κάναμε ειδική νομοθεσία τότε στην Κύπρο για τις αμβλώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία που μας προσφέρατε ότι έχει σαφή ε, θέση η Κύπρος. Και τώρα η κυρία, η κυρία Κλοντέτ Ποτιτζίτζι, λέει ο πρόεδρος. It's Buttigieg, αλλά εντάξει. <laughs> Καλημέρα σας. Είμαι από τη Μάλτα και όπως ε, θα γνωρίζετε πολύ καλά η χώρα μου για πολύ καιρό ήταν ε, χώρα ε, μεταναστών. Τώρα έγινε χώρα ε, διέλευσης και αυτή τη στιγμή έχει γίνει και μια χώρα ε, στην οποία δεν επιθυμούν να έρθουν ε, οι ε, μετανάστες. Αρκετοί πρόσφυγες που έρχονται στη χώρα μας δεν θέλουν να μείνουν εκεί, θέλουν να πάνε αλλού. Αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα στην Ευρώπη συνέβαινε όμως στη χώρα μου για πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι χάθηκε πολλής χρόνος. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρα πολλά πράγματα ως δίδαγμα για την πραγματικότητα της χώρας μου, της Ιταλίας, της Ελλάδος και μάλιστα της Ελλάδας που συνεχίζει να υποδέχεται πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρώτον, τι κάνουμε στη χώρα καταγωγής ε, αυτών των γυναικών και παιδιών και των υπολείπων προσφύγων. Νομίζω δεν γίνονται αρκετά. Πάντα προσπαθούμε ε, εμβαλωματικά να λύσουμε το πρόβλημα όταν προκύπτει. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε λίγο καλύτερα στις χώρες καταγωγής. Η Συρία είναι περίπλοκη, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, περιπτώσεις, τις οποίες νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Κάτι άλλο. Τον Ιόνιο του 2014 ήμουνα σε μια διάσκεψη για τη σεξουαλική βία και τις συγκρούσεις στο Λονδίνο. Έγιναν πολλά εκεί, πολλές χώρες ε, προσυπέγραψαν ε, το Διεθνές Πρωτόκολλο για την Προστασία των Γυναικών από την ε, σεξουαλική βία σε περίοδο σειράξεων, όπως είπε και η κυρία Κιέγγε προηγουμένως. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν βλέπουμε γυναίκες έγκυες σε ένα πλοιάριο θα πρέπει να τους ρωτήσουμε ήθελαν αυτή την εγκυμοσύνη, πώς προέκυψε, ε, αποτελεί αυτό εισιτήριο για αυτούς τους άντρες ε, για να μπορέσουν να τους αφήσουν να έρθουν στη χώρα μας. Ε, πρόκειται για πολύ σοβαρά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσέκρετσι από την Αλβανία είναι η τελευταία ομιλητρία μας. Ist die Dame nicht mehr im... Μήπως έχει βγει από την αίθουσα, κυρία Τσερκέζη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όπως και οι συνάδελφος από την Αλβανία. Θέλω να μιλήσω για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες που φεύγουν από την Αλβανία. 20% είναι γυναίκες και παιδιά. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και τραυματικές εμπειρίες, εκ των οποίων η μία είναι και η απουσία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Πρέπει η Ευρώπη να βοηθήσει, να καταργήσει τους φραγμούς και τα σύνορα, να τις βοηθήσει να φτάσουν σε σταθμούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσοκομεία Πολλές είναι οι Αλβανίδες οι οποίες έφυγαν από την πατρίδα τους έγκυες ούσες. Χρειάζονται υποστήριξη. Χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια για τις γυναίκες αυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλιότερα θα έβγαν οι άντρε ω πρόσφυγε από την Αλβανία, αφήνοντα πίσω τι οικογένειέ του στη χώρα. Πρέπει να εξασφαλιστούν περισσότερε ευκαιρίε για αυτού ώστε να ξαναβρεθούν μαζί οι οικογένειες. Ζητούμε λοιπόν υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε να σταματήσει η γραφειοκρατία και να βελτιωθούν οι διαδικασίες ώστε να μπορέσουν να βρεθούν κοντά οι οικογένειες. Η Πρόεδρος νομίζω ότι μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο που είχαμε σε θέση μας πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, για τις τοποθετήσεις σας είχα άχαρο καθήκον ε, να πρέπει πάντα να σας κόβω το λόγο. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ε, ήταν γιατί δεν ήθελα να σας αφήσω να μιλήσετε, αλλά γιατί έπρεπε να δώσουμε το χρονικό περιθώριο σε όλες τις ομιλητρίες. Στις 11 πρέπει να ξεκινήσει η Ολομέλεια για να μιλήσουμε για τις εργασίες του κάθε workshop. Έχετε εδώ τη δυνατότητα να πάρετε ένα καφέ έξω από την πόρτα της αίθουσας, εάν το θέλετε. Σας παρακαλώ πίσω να είσαστε στις 11 ακριβώς για να αφήσουμε ε, το χρόνο για την Ολομέλεια. Για δε τις απαντήσεις από τους, ειδικές, από τους ειδικούς μας ήταν ε, νομίζω προτιμότερο να αναπτύξετε διμερώς αυτές τις επαφές ε, για να λάβετε τις απαντήσεις σας κατά τρόπο πιο αποδοτικό και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση των μας με την Ολομέλεια. Ευχαριστώ.